Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Καθίστε. Περιμένουμε την κυρία Μπούλτς. Στο μεταξύ, θα ήθελα να διορθώσω ένα σφάλμα που έγινε σήμερα το πρωί. Όταν σήμερα το πρωί στις 10 σας είπα ότι είχε 40 βαθμούς έξω. Όχι, δεν είχε 40 βαθμούς, αλλά 30. Δεν θέλω fake news να κυκλοφορούν ε, στην Επιτροπή μου, έτσι διορθώνω. Τώρα όμως έχει 36 βαθμούς, όχι 40, 36. Έτσι, διορθώνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σας παρακαλώ να υποδεχτούμε εδώ για το επόμενο σημείο μας την Επίτροπο, την κυρία Μπούλτς, για την παρουσίασή της. Φτάνει. Jesus, what an Mes chers collègues, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μια μισή ώρα θα περάσουμε μαζί με την κυρία Μπούλς για να μάθουμε ε, τι ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιος είναι ο επόμενος χάρτης πορείας της κλπ. Πραγματικά θα φροντίσουμε να μάθουμε ποια είναι τα τελευταία αποτελέσματα του Συμβουλίου Μεταφορών και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και τα κείμενα τα οποία περιμένουν να τα προχωρήσει η Επιτροπή. Ξέρω πόσο πολύ ενθουσιάζεται με τις μεταφορές η Βιολέτα. Θα της, θα δώσω 10 λεπτά για την αρχική της παρουσίαση. Άντε 12. Και μετά, όπως και πριν, θα έχουμε ένα πρώτο γύρο με ερωτήσει από τους συντονιστέ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ξέρετε, ένα λεπτό ο καθένα για την ερώτησή του και μετά θα κάνουμε και νέα γύρο για τους υπόλοιπου ευρωβουλευτές, εφόσον έχουν κάποια ερώτηση, πάλι για ένα λεπτό θα μπορούν να ρωτήσουν την Επίτροπο. Εκτός από τους συντονιστές είπαμε θα έχουμε δεύτερο γύρο και όποιος θέλει να πάρει το λόγο να μας το πει να του σημειώσουμε, έτσι. Ωραία, έτοιμοι. Παρακαλώ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και τώρα, σήμερα, νόμιζα ότι όλοι είχαν ήδη φύγει διακοπές, αλλά βλέπω ότι εξακολουθείτε να εργάζεστε εσείς. Και χαίρομαι που βλέπω εδώ κάποια γνωστά πρόσωπα, όχι όμως και τόσο πολλά στην πραγματικότητα. Ε, ξέρω όμως ότι πιο έμπειροι παραμένουν και σίγουρα θα βοηθήσουν με τη δικιά τους εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα τελευταία πέντε χρόνια, θα την περάσω και στους νέους. Χαίρομαι όμως που βλέπω και καινούργια πρόσωπα εδώ. Νέους ευρωβουλευτές. Εσείς είσαστε εδώ για να αμφισβητήσετε τα πάντα, για να μας ρωτήσετε, για να μας βοηθήσετε να ανανοθούμε. Θα συνεργαστούμε λοιπόν μαζί για να ετοιμάσουμε το μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών τα επόμενα πέντε χρόνια. Φυσικά και είμαι στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε τώρα στο τέλος της δικιάς μου εντολής και να ολοκληρώσουμε κάποιους από τους φακέλους που παραμένουν σε εκκρεμότητα αλλά που είναι ζωτική σημασία για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών μεταφορών. Πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή σας σίγουρα είναι μία από τις πιο δραστήριες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κάθε δύο μήνες έπρεπε να έρθω εδώ για νέα ακρόαση. Και κάθε φορά που ερχόμουν εδώ στο Ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο οι συζητήσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, και επικεντρωνόντουσαν ε, πολύ συγκεκριμένα και πραγματικά στα πιο βασικά ζητήματα για τα οποία θα έπρεπε μαζί να βρούμε λύσεις. Είναι λοιπόν προνόμιο για μένα και ιδιαίτερη χαρά που συνεργάζομαι με όλους εσάς. Όμως δεν έχουμε τελειώσει. Εσείς τώρα ξεκινάτε σε μια περίοδο που στην πραγματικότητα επαρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο δυναμισμό. Θα αναφέρω κάποια θέματα μόνο. Έχουμε την κλιματική αλλαγή εννοείται και τις επιπτώσεις ε, στο κλίμα. Πριν από τέσσερα χρόνια αρχίσαμε να εντοπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα όμως δεν ήταν ε, μέσα σε κάθε πολιτική, σήμερα ναι. Και ξέρουμε ότι οι μεταφορές είναι υπεύθυνε για το 24% όλων των εκπομπών, αλλά και για άλλου είδους ρήπανση στον αέρα. Η ευθύνη των μεταφορών λοιπόν είναι μεγάλη, οπότε σας παρακαλώ πολύ να είσαστε ρεαλιστές και να φροντίσετε να βοηθήσετε όλες τις πλευρές ώστε να φέρουν αποτελέσματα Ξέρουμε ποιο είναι το όραμά μα για το 2050 και πιστεύω ότι είναι εφικτό και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η ψηφιοποίηση επίση αποτελεί μια μεγάλη τάση με την οποία έχουμε ήδη ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να κάνουμε με περισσότερες εναλλακτικέ λύσεις για νέες παρεμβάσεις από την πλευρά μας, ώστε να υπάρχει ισότητα, να υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός στην εσωτερική μας αγορά, αλλά και παγκοσμίω. Έπειτα έχουμε και απειλές για την ασφάλεια. Αυτές δεν εξαφανίζονται ποτέ. Τα θέματα της ασφάλειας, δηλαδή και της προστασίας των πολιτών, αποτελεί την βασική αξία των μεταφορών μας. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Οι μεταφορές πρέπει να είναι ασφαλείς. Έπειτα, περιορισμοί στην αγορά. Και όχι μόνο. Και αυτό και άλλα ζητήματα θα τα βρείτε μπροστά σα σε αυτή τη θητεία. Ξέρω όμω ποια είναι η φιλοσοφία τη Επιτροπή Μεταφορών και ξέρω ότι ό,τι και να γίνει, εσεί θα βρείτε τον τρόπο να το αντιμετωπίσετε. Και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα έχετε έναν εξαιρετικό επίτροπο, ο οποίο θα συνεργαστεί πολύ καλά μαζί σα. Όλε αυτέ οι προκλήσει λοιπόν, αλλά και ευκαιρίε που έχουμε μπροστά μα και που πρέπει να αντιμετωπιστούν, είναι πολλές. Εμείς όλα αυτά προσπαθούμε να τα βάλουμε κάτω από ένα καπέλο. Και σας ζητώ να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έρχονται διάφορα πολιτικά μηνύματα. Και υπάρχει και το όραμα 0, το τριπλό 0, που είναι 0 ρήπανση, 0 δυστυχήματα στους δρόμους ε, αλλού, και 0 γραφειοκρατία κυρίως χαρτί, να μην χρησιμοποιούμε χαρτί. Και ούτε να επιβάλλουμε υπερβολική γραφειοκρατία στους επιβάτες. Αυτά είναι τα 3 μηδέν. Αλλά χρειάζονται πολλά βήματα προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτά τα 3 μηδέν. Στην τελευταία θητεία που συνεργάστηκα μαζί σας, μπορέσαμε να περάσουμε 49 νομοθετικούς φακέλους που σημαίνει ότι ήμασταν πάνω-πάνω μεταξύ των διαφόρων χαρτοφυλακίων της προηγούμενης θητείας. Πετύχαμε σε 33, που είναι τεράστιο πίτευμα και σας ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που βοηθήσατε για να τα καταφέρουμε. Όμως παραμένουν 16 προτάσεις ακόμα σε κραμότητα και βασίζομαι στη δικιά σας την ε, βοήθεια και τη στήριξη για να προχωρήσουμε και σε αυτούς τους φακέλους και ελπίζω να τα καταφέρω στην εντολή μου να το κάνω αυτό μαζί σας. Επίσης, ξεκινήσαμε διάφορες διαπραγματεύσεις όσον αφορά ε, διεθνείς συμφωνίες μεταφορών και ε, παράγωγο δίκαιο, παράγωγες νομοθετικές πράξεις. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ σε κάποιους φακέλους που είναι σε κρεμότητα και κυρίως τους δύο που θεωρούμε ότι είναι οι πιο επίγοντες. Πρώτον, έχουμε τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, νούμερο 2. Και στη συνέχεια έχουμε και το πακέτο κινητικότητας 1. Έχουμε επίσης τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που έχουν προχωρήσει πολύ, κυρίως για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη 2, που διαμορφώθηκε μερικώς μια συμφωνία τον Απρίλιο. Ελπίζω πάντως ότι μπορώ να βασιστώ σε εσά για να προχωρήσουμε περισσότερο. Δεν μπορώ να τονίσω ποτέ αρκετά πόσο μεγάλη σημασία έχει να συνεχίσουμε να έχουμε επενδύσεις στις μεταφορές στην Ευρώπη. Αν σταματήσουν οι επενδύσεις τελείωσε. Αν δεν έχουμε επενδύσει στις μεταφορές, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να βοηθήσετε και να ενημερώνετε και στις χώρες σας ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα μεταφορών. Για παράδειγμα, εμείς ε, κάναμε πολλές εκκλήσεις τα τελευταία 4,5 χρόνια. Κάθε φορά, από δύο μέχρι και 7 φορές, ε, καταφέραμε να κινητοποιήσουμε ποσά παραπάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έπειτα, το πακέτο κινητικότητα. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πριν από δύο χρόνια το πακέτο αυτό για την καλή λειτουργία τη αγορά οδικών μεταφορών και για να υπάρχουν και καλύτερε συνθήκε εργασία για του οδηγού. Πέρασε ο καιρό, η κατάσταση όμω επιτόπου δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Αντίθετα, μάλιστα, θα έλεγα, επιδεινώνεται. Αυτό σημαίνει ότι το πακέτο δεν προχώρησε και οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Τελικά, τελικά κάποιος κερδίζει, κάποιος φαίνεται να χάνει, δεν χάνει όμως, η δημοκρατία κερδίζει. Υπάρχει όμως περιθώριο ακόμα για βελτίωση, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που η Φιλανδική Προεδρία με διαβεβαίωσε ότι και αυτοί είναι έτοιμοι να αναλάβουν αμέσως μόλις εσείς είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουν τριμερή διάλογο μαζί σας. Και όπως σας είπα και πριν, είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε παρετέρω το πακέτο για να το προσαρμόσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κάποιες τρίτες περιφέρειες. Χρειάζεται όμως το πακέτο. 60% του διοικητικού άχθους φτάνει για να μας πείσει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να προσελκύουμε νέους. Γιατί βλέπετε ότι το επάγγελμα αυτό δεν έχει νέους, δεν έχουμε οδηγούς. Και δεν έχουμε οδηγούς όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά εξαιτία των συνθήκων κάτω από τις οποίες εργάζονται. Εξαιτία των συνθήκων εργασίας τους. Οπότε, σας παρακαλώ πολύ, να προχωρήσουμε, γιατί είναι κάτι που χρειάζεται ο κόσμο το χρειαζόμαστε όλοι. Έπειτα, συνδυασμένε μεταφορέ. Ε, πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει, όπω είπαμε, για το πακέτο κινητικότητα αριθμό 1. Αλλά έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για τι συνδυασμένε μεταφορέ. Το έχει πει το Συμβούλιο. Είναι και αυτή δηλαδή μια προθεσμία που έχουμε μπροστά μα. Γιατί έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό και πρέπει αυτό το πρώτο βήμα να το ολοκληρώσουμε. Όπως ξέρετε δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεταχειριστεί τις ε, συνδυασμένες μεταφορές. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε στο χειρότερο πακέτο και στο κακό πλαίσιο που έχουμε σήμερα, άρα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ για να το διορθώσουμε και να εκπονήσουμε την κατάλληλη νομοθεσία που να λειτουργεί ως κίνητρο και να βοηθάει και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι το EFTI. Τον Ιούνιο, στη συνάντηση του Συμβουλίου, ενέκρινε μια γενική προσέγγιση η, η Υπουργή Μεταφορών όσον αφορά τις ε, ηλεκτρονικές πληροφορίες μεταφορών. Είναι ένας ε, φάκελος ο οποίος ελπίζουμε να ολοκληρωθεί υπό Φιλανδική Προεδρία. Ε, χτες συναντήθηκα μαζί τους και σήμερα νομίζω και υποσχέθηκαν ότι θα το προχωρήσουν. Και γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό, γιατί έτσι οι πληροφορίες για τις εμπορικές μεταφορές θα είναι ψηφιακές και έτσι θα μειωθεί το κόστος κατά 22 με 27 εκατομμύρια το 2040. Ελπίζω αυτό από μόνο του να βοηθάει να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρώσουμε. Τον Ιούνιο επίσης το Συμβούλιο συζήτησε και έκθεση πρόοδου για άλλους φακέλους σημαντικούς και θέλω να πιστήσω την προσοχή σας αυτούς γιατί ελπίζω ότι θα τους κοιτάξει η Φιλανδική Προεδρία επίσης. Πρώτον, γιατί είναι Ευρωβινιέτα. Χρειάζεται επίσης το streamlining με απλοποιημένες διαδικασίες όσον αφορά τις υποδομές των διευρωπαϊκών δικτύων. Να μπορούμε να έχουμε τα έγγραφα που χρειάζονται και να ετοιμάσουμε ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορέσουμε και να επιταχύνουμε τις διοικητικές αυτές διαδικασίες για τα τέντη, έτσι ώστε όλοι οι διάδρομοι να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και να μπορέσουμε έτσι να προσφέρουμε συνολικά δίκτυα το 2050. Έπειτα για τα ενοικιαζόμενα οχήματα, να διευκρίνουμε την ε, ενοικίαση ε, ελαφρών και βαρέων οχημάτων σε άλλες χώρες μέλη. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί υπάρχουν εδώ πολλές προκλήσεις στην αγορά όσον αφορά τα οχήματα αυτά. Η αντιμετώπιση όμως πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Και τέλος υπάρχουν και τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων. Και εδώ πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες. Η Φιλανδική Προεδρία είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί και με αυτό το θέμα και να φέρει αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω λίγα λόγια για την Ευρωβινιέτα. Διότι μερικές φορές ακούμε διαφορετικές ερμηνείες στα μέσα ενημέρωσης για το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε να πετύχουμε με αυτό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πιέζουν τις μεταφορές να μειώσουν τις επιπτώσεις των μεταφορών στο περιβάλλον. Και η Ευρωβινιέτα μας βοηθάει οι ρηπαίνοντες να βοηθήσουν. Δηλαδή αυτός που ρηπαίνει να πληρώνει για την ρήπανση που προκαλεί και για τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα το θυμόσαστε. Τέσσερα χρόνια μας πήρε να έχουμε μία έκθεση με την εξωτερήκευση του κόστους κλπ. Κοιτάξτε την έκθεση αυτή, αξίζει τον κόπο. Και νομίζω ότι από αυτή την πρόταση θα έχουμε και πολλές νέες προτάσεις. Το λέω πάντως ξανά ενώπιόν σας και να το πείτε στους πολίτες σας ότι χαιρόμαστε που πραγματικά κάνουμε βήματα προς τα μπρος για να βρούμε λύσεις για αυτούς που κυκλοφορούν καθημερινά στους αυτοκινητοδρόμους. Πρέπει να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Και δύο λόγια για την αεροπορία. Αεροπορικές μεταφορές. Φυσικά και θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο μας για διάφορους φακέλους. Ξέρετε ότι σταματήσαμε ενώ είχαμε διαπραγματευτεί διάφορες συμφωνίες που συνεισφέρουν σε πραγματική βελτίωση της σύνδεσης στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμως να τους θέσουμε και σε εφαρμογή. Έχουμε κολλήσει. Έχουμε τη διαχείριση των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ζήτημα του Γιβραλτάρ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την απογοήτευσή μου. Χάνουμε 2,8 δισεκατομμύρια ετησίως απλώς και μόνο επειδή δεν μπορούμε να έχουμε συνολικές συμφωνίες. Και δεν μιλάω εδώ μόνο για το θέμα της συμφόρησης, που όλοι θα το έχετε διαπιστώσει φέτος. Δεν μπορούμε όμως να βελτιώσουμε τα πράγματα, γιατί χρειαζόμαστε ομοφωνία στο Συμβούλιο και το ζήτημα του Γιβραλτάρ δεν έχει λυθεί ακόμα και δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τι μεταφορέ. είναι διπλωματικό το ζήτημα όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια διπλωματική διαφωνία και πρέπει να λυθεί σε επίπεδο επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Βοηθήστε μας λοιπόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να βρεθεί δηλαδή μια λύση σε αυτό. Νομίζω ότι εξαντλήθηκε ο χρόνος μου. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Το μόνο που θέλω να πω τελειώνοντας είναι ότι το γεγονός ότι είναι τόσο γεμάτη η αίθουσα αυτή σήμερα δείχνει ότι οι μεταφορές είναι κάτι που έχει μπει και πάλι στο αυλάκι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη θητεία σας και ό,τι καλύτερο και τις ευρωπαϊκές μεταφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ, Βιολέτα, που μας υπενθύμισε τους μεγάλους στόχους με τα ίδια θέματα πάντα. Πακέτο κινητικότητα, συνδικές εργασίες ε, οδηγών. Το Συμβούλιο έχει μία θέση, αυτό πρέπει να θυμίσουμε. Μία θέση, το Κοινοβούλιο έχει μία θέση, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ε, το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων θα καθοριστεί στην επόμενη συνάντηση με τους συντονιστές. Σας θυμίζω ότι αλλάξαμε. Κάποιοι βουλευτές δεν είναι πλέον βουλευτές. Χρειάστηκε να αλλάξει και ο εισηγητής που δεν θα καθυστερήσει πολύ τη διαδικασία. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που είπατε κύριε Πίτροπε, είναι ότι δεν μπορούμε να χάσουμε περαιτέρω χρόνο για κείμενα που είναι στα συρτάρια και όπου υπάρχει ήδη θέση του Κοινοβουλίου. Ευρωβινιέτα. Ένα εργαλείο δράσης κατά της αλλαγής του κλίματος. Αυτό πρέπει να προχωρήσει για να, να, για να πάρει μπρο ο κλάδος, ιδίως των εμπορευματικών μεταφορών. Πρέπει να ξαναπάμε τα εμπορεύματα στο Σιβιόδρομο. Τουρισμός, ένα θέμα που δεν σχολιάσαμε πολύ. Αυτή είναι λογική όμως του βιώσιμου τουρισμού, όχι τα τεράστια κουρασγερόπλια που φτάνουν στη Βενετία και δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πλεούμενα νησιά. Έτσι, Ιζαμπέλα. Κατόπιν, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι νέο, να εφεύρουμε κάτι νέο, να λάβουμε υπόψη κλάδους που δεν είναι συνήθεις ε, στις συζητήσεις. Η, η ναυτιλία έχει επιπτώσεις στο, στην ρήπανση, στο κλίμα. Αερομεταφορές Θέλουμε ένα πακέτο αερομεταφορές. Κοινωνική, ένα κοινωνικό πακέτο. Δεν μπορεί να δουλεύουν αεροσυνοδοί και πιλότοι κατά από άθλιες συνθήκε. Ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και την περιβαλλοντική διάσταση. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ο κλάδος. Μια τελευταία παρατήρηση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το είπα το πρωί και δεν θα αλλάξω θέση δικαιώματα των επιβατών. Πρέπει να διαπραγματευτούμε. Έγινε λόγος για τη μελέτη για την ε, διαλειτουργικότητα. Αυτό τι σημαίνει. Να προχωρήσουμε σε δράσεις που δεν είναι ακριβά, ακριβές. Το ποδήλατο στο τρένο, για παράδειγμα. Υπάρχουν δικαιώματα καταναλωτών. Το, θέλει, δεν μπορεί να έχουμε μία-δύο θέσεις για ποδήλατα σε κάθε τρένο ή α το καταργήσει το Συμβούλιο άμα θέλει. Κατόπιν δεν μιλήσατε και αυτό ήταν ένα μεγάλο κομμάτι των διαπραγματεύσεων με τους παλιού. το Brexit. Έρχεται, μπροστά μας είναι. Εμείς κάναμε αυτό το πλέγμα ασφαλείας για τις αερομεταφορές και τις οδικές μεταφορέ, αλλά αν δεν υπάρξει συμφωνία θα παραλύσουν τα πάντα. Στις αεροπορικές μεταφορές, στις σιδηροδρομικές, στις μεταφορές, στις εμπορευματικέ. Τι κάνει η Επιτροπή. Σκέφτεται τις, τα ενδεχόμενα. Άλλο θέμα, προπολογισμό. Πρέπει να κρατήσουμε τον προπολογισμό της Επιτροπής Μεταφορών. Πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε το ποσό αλλά και να επαναπροσανατολίσουμε τον προπολογισμό. Οι πολίτες περιμένουν συγκεκριμένα πράγματα από εμά. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο και μιλώ συγκεκριμένα. Εγώ είπα τα συγκεκριμένα πράγματα, περιμένω και από εσά να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Για ένα λεπτό, κύριε Τέλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καλησπέρα σας κυρία Επίτροπε εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας και για τη γενική διεύθυνση MOVE. Ε, πετύχατε αρκετά πράγματα παρότι το περιβάλλον πρέπει να πω ότι δεν ήταν η πρώτη σας προτεραιότητα. Η Επιτροπή Μεταφορών αναγκάστηκε όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. και μην το παρεξηγήσετε, πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα, όμως δεν μπορούν είναι το μόνο που θα μας απασχολεί. Γι' αυτό ας συνεργαστούμε με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ε, για τα θέματα αυτά, ε, γιατί μας ενδιαφέρουν τα θέματα της κινητικότητας και του τουρισμού. Υπάρχουν σημαντικά θέματα όπως τα δικαιώματα των πολιτών. Εκεί δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος. Για το Γιβραλτάρ και εκεί ε, υπολείπονται ακόμα αρκετά. προσπαθήσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Έχω κατά νου ότι Βεβαίως ε, έχουμε μία πρόεδρο που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το πρασίνισμα του τομέα των μεταφορών, γιατί εκπροσωπεί τους πράσινους. Εγώ θα ήθελα ε, στη μελλοντική δουλειά μας να βρούμε μια καλύτερη ισορροπημένη προσέγγιση. Υπενθυμίζω ωστόσο ότι η εντολή της νέας Προέδρου της Επιτροπής έχει ως προτεραιότητα το κλίμα, το είπε. Άρα χαίρο που η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΛΚ, πιέζει για να υπογραμμιστεί τη σημασία του κλίματος. Κύριε Αρτώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόση ώρα έχω. Ε, ένα λεπτό, μόνο ένα λεπτό. Άρα τι να κάνω σε ένα λεπτό, δεν μπορώ να ρωτήσω τίποτα. Τέλος πάντων. Ε, κύριε Μπούλτς, ε, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου εκ μέρους των σοσιαλιστών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Νομίζω ότι στο τέλος γίναμε μια πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, προσπάθειές σας. Έχω πολλές ερωτήσεις και έχω να ασκήσω και κριτική. Ξεκινώ πρώτα με την κριτική. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα τέλη διοδίων και θέλω να πω ότι και εσείς και ο κύριος Γιούγκερ ε, δεν παίξατε και πολύ καλό ρόλο στο θέμα αυτό. Αυτή είναι η κριτική μου. Ερώτηση τώρα. Ε, το θέμα πολύ προβληματικό που αφορά τη Βαβαρία και την Αυστρία. Γνωρίζετε ότι τα φορτηγά ε, που διασχίζουν της Άλπης, ε, το Μπρένερο, ε, είναι υπό διαπραγμάτευση. Γνωρίζω ότι έχει επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το άλλο που θέλω να σου είναι για τα δίκτυα TEN-T, TEN-10. Ε, κάναμε πάρα πολλά. Πρόκειται να εφαρμοστεί το πρώτο. Ε, ημουν εισηγητής 21-22. Πρόκειται για το, πρώτο πρόγραμμα αναθεώρησης. Έχετε να μα πείτε κάτι συγκεκριμένο από αυτού. Και το δεύτερο, 11,3 δις ευρώ. Ε, αυτό δεν αρκεί. Μήπως υπάρχει κάτι για να αυξήσουμε αυτό το ποσό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπόσας Δίας. Ισπανικά θα σας τα πω. Η παρέμβαση της ομάδας μου δεν αφορά στο να σας θέσει ερωτήσεις αλλά να σας ευχαριστήσει απλώς για τη δέσμευση και την αφοσίωσή σας στην, στο φωτοφυλάκιο αυτό για τις προσπάθειες και αφοσίωση λέω που διαπιστώσαμε ανα πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας σας και να σας πω ότι η ομάδα μας που είναι η τρίτη στην, ε, στο Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχουμε όσες περισσότερες συμφωνίες γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες του Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευαίσθητοι φάκελοι, εν κάποιοι είναι ήδη επιτάπητος, άλλοι θα έρθουν. Η δέσμευσή μας ως τρίτη ομάδα στο Κοινοβούλιο είναι να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Και για να μην λέτε ότι θα κάνουμε καμία ερώτηση, θα έλεγα από τα χρόνια σας πείτε μας τι σας ικανοποιεί περισσότερα τι πιστεύετε ότι, πώς πιστεύετε ότι περισσότερο συμβάλλατε, ποιες είναι οι, αυτά που πετύχατε σαν επίτροπος. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Monsieur la parole est à vous. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα κύριε Επίτροπε να σας ε, καλωσορίσω ε, και θέλω να σας πω ότι έχει έρθει πια η χρονική στιγμή για μας για να σκεφτούμε τι ακριβώς συνέβη τα τελευταία πέντε χρόνια σε επίπεδο Επιτροπής. Ε, εξετάζοντας λοιπόν αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ε, θερμοκρασίες ρεκόρ. Νομίζω ήδη έχουμε 41 βαθμούς εχθές στη Γαλλία. Αύριο το πρωί στο Ηνωμένο Βασίλειο η θερμοκρασία θα ξεπεράσει το 38,5 και τώρα είναι 36 βαθμοί εδώ έξω στις Βρυξέλλες σήμερα. Παράλληλα ε, την τελευταία ώρα είδα ότι η ήλιο μας ε, επισήμανε ότι έχει αλλάξει, έχει χαλάσει η ποιότητα του του αέρα στι Βρυξέλλε. δεν μας λέει να μην οδηγούμε να προστατευτούν κυρίω τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Ε, τα τελευταία πέντε χρόνια πιστεύετε ότι κάνατε αρκετά για να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή ή πιο συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσετε το θέμα ε, τη ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Γιατί γνωρίζουμε ότι το εξωτερικό κόστο των μεταφορών ε, κυμαίνεται περίπου στο 1 δι ευρώ σε τήσια διαβάσει αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος και πιστεύω ότι είναι και ένα θέμα ιδεολογικό. Και αυτό το θέμα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκοντας ε, την επίτευξη της ε, κοινή αγοράς και τη διευκόλυνση των ταξιδιών, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στο να εκπέπονται περισσότερες εκπομπές ε, στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε από αυτού κατά τη διάρκεια το τι ακριβώς συνέβη κατά τη της περίοδου ως επίτροπος. Αν μπορείτε να τηρήσετε το χρόνο θα ήταν ε, χρήσιμο για όλους μας. Ο κύριος Έντερ έχει το λόγο. Θα σας μιλήσω γερμανικά. Εγώ ως Αυστριακός ε, Ευρωβουλευτής θέλω να σας πω ότι όλη η συζήτηση για την Ευρωβινιέτα είναι πολύ σημαντική για μας ε, γιατί το σύστημα ε, είναι λιπές και εγώ πιστεύω ότι ένα εύρυθμα λειτουργούν σύστημα δεν θα πρέπει να αλλάζει. Ε, όσον αφορά αυτή την οδηγία, εμείς δεν θέλουμε να προκύψει επιπρόσθετο κόστος και για επιχειρήσεις, αλλά και για ιδιώτες, για πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία Επίτροπε, θέλω να σας ερωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα κείμενο που το ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Εκεί εξαιρούνται τα γιοταχή. Προτίθεστε να τα ξανασυμπεριλάβετε και αν ναι, από πότε και ποια θα είναι η εφαρμογή αυτής της πρότασης. Και έχω και μία δεύτερη ερώτηση σχετικά με τα διόδια. Εμείς ε, προτείνουμε να ε, μην τοποθετηθούν εκ των υστέρων ε, ταχογράφοι. Τι ακριβώς πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή έχει βελτιωθεί η τεχνολογία, μήπως σκέφτεται κάποια άλλη τεχνολογία, παραδείγματο χάρη να χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα. Μήπως προβλέπετε μία app, μία εφαρμογή που θα αντικαταστήσει τους ταχογράφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να πω σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη δουλειά σας για αυτά τα πέντε χρόνια και Ακόμα και αν είχαμε πολύ καλή συνεργασία, σε κάποια θέματα είχαμε και διαφορετικές απόψεις, ε, όπως παραδείγματος χάρη στο πακέτο της ε, κινητικότητας. Θα ήθελα να συνδυάσουμε την ε, τρέχουσα μορφή του πακέτου κινητικότητας με άλλες δυνατότητες. Εσείς είχατε για το 2050 όνειρα να μην υπάρχουν καθόλου εκπομπές, ίσως το 2050 να μην υπάρχουν και καθόλου οδηγοί φορτηγών. Όμως με βάση το ε, πακέτο της κινητικότητας ε, ε, τα φορτηγά θα μετακινούνται χωρίς οδηγό, θα μετακινούνται από τη Λετωνία μέχρι τη Γερμανία και αυτά θα περνάνε στους δρόμους, ε, δεν θα έχουμε όμως τους οδηγούς. Ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει κάπως να τα διαχωρίσουμε όλα αυτά. Και επίσης ε, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί το τι θα γίνει το πακέτο κινητικότητας. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβρη. Η κυρία Κουντουρά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για τις πρωτοβουλίες σας και για το έργο σας τα, τέσσερα τελευταία, τα πέντε τελευταία χρόνια. Ε, μιλήσατε για το πακέτο κινητικότητας, το οποίο όντω έχει πολύ μεγάλη σημασία και θεωρούμε και εμείς ότι είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν οι μακροχρόνιες να μην πάνε χαμένες είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αφορά ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους Ευρωπαίους οδηγούς και σημαίνει παράλληλα και αυξημένη ασφάλεια. Γι' αυτό πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι τριμερείς ε, διάλογοι και αυτός ο συμβιβασμός που πετύχαμε ε, να συνεχίσει έτσι ώστε να μην καθυστερήσουμε και χαίρομαι που δεσμεύεστε κι εσείς για να προχωρήσει. Η κλιματική αλλαγή ε, είναι προτεραιότητα όπως υπόθηκε και από εσάς αλλά και από τους προηγούμενους ομιλητές. Και πάντα όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Μία ερώτηση λοιπόν που θα ήθελα να σας κάνω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση για τις πράσινες μεταφορές ε, που πρέπει να βάζουμε ε, επίκεντρο τον άνθρωπο και το κοινωνικό στοιχείο. Εάν επιβαρύνουμε τις μεταφορές των αγαθών και των επιβατών δεν θα αποκλείσουμε τα φτωχότερα ε, στρώματα. Μήπως παράλληλα χρειάζεται να πάρουμε και αντισταθμιστικά μέτρα για τους πιο αδύναμους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Κουντούρα. Κυρία Επίτροπε, πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Καρίμα. πολλές ερωτήσεις, να δώσω και κάποιες εξηγήσεις. Η Καρίμα έθεσε όλο το πλαίσιο που πρέπει να συζητήσουμε, αλλά και οι επιπλέον ερωτήσεις ήταν ε, πολύ σαφείς. Γιβραλτάρ, κύριε Τάλερ, πρώτη εγώ θα χοροπηδούσα από τη χαρά μου αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω την πρόταση που χρησιμοποιούμε σε άλλους φακέλους για να λύσουμε για να αφήσουμε την, ε, την περίπτωση του Γιβραλτάρ απ' έξω. Δυστυχώς το Brexit μπλόκαρε τα πάντα. Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα ή οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν να απελευθερώσουν να, το, την αεροπορική, τις αεροπορικές μεταφορές από την παγίδα τους πάνω από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται. Αλλά δεν έχουμε εξουσία πάνω σε αυτό. Πάντως, πιστέψτε με, πρώτη εγώ θα χοροπηδούσα από τη χαρά μου. Περιμένουμε. Είμαστε stand-by και έτοιμοι να πηδήξουμε. Για την πράσινη θεματολογία, το Green Agenda, πολλοί το ανέφεραν. Όταν ήρθα, δεν ανησυχούσαμε πάρα πολύ για την ρήπανση ακόμα. Όντως, πριν από πέντε χρόνια η κατάσταση ήταν διαφορετική από τώρα. Από την πρώτη όμως ημέρα ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που είχαμε στη διάθεσή μας για να παροτρύνουμε ένα επενδύσεις στην, στο πρασίνισμα των μεταφορών. 80% των, των, των επενδύσεων της προηγούμενης περίοδου το χρησιμοποίησαμε για τις ιδεοδομικές μεταφορές και τις εσωτερικές πλωτές οδούς, πράσινα, πράσινα μέσα, πράσινες μορφές μεταφοράς. Το ίδιο ισχύει και την επόμενη χρηματοοικονομική περίοδο. Εξασφαλίσαμε ότι οι περισσότερες επενδύσεις θα στραφούν στην πράσινη ατζέντα. Συνεχίζουμε λοιπόν να πιέζουμε προς αυτό. Είμαστε οι πρώτοι που είχαμε δηλώσει ε, μηδενικές εκπομπές το 2050. Χαίρομαι που αυτό το υιοθετούν και άλλα χαρτοφυλάκια. Το ξέρουμε για δύο λόγους. Πρώτον, θέλαμε να ακολουθήσουμε την συνολική στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης που λέει ότι πρέπει να, να αναζητήσουμε πιο κατανεμημένες πηγές τροφοδοσίες, ε, ενέργεια και, να, και περισσότερο πρά, πράσινες μορφές ενέργειας από τις οποίες δεν είμαστε εξωτερικά εξαρτημένες. Γι' αυτό προχωρούμε τώρα σε εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, ιδίω στην ε, διαμόρφωση των υποδομών που θα επιτρέπουν, που θα δίνουν πρόσβαση στους χρήστες των μεταφορικών μέσων σε αυτές τις εναλλακτικέ μορφές ε, καυσίμων. Επίσης, ε, είχαμε τις ε, φιλόδοξες, τους φιλόδοξους στόχους για τα όρια εκπομπών των αυτοκίνητων, ιδίως των ΙΟΤΑΧΗ. Μπορεί να έχουμε και πολύ πιο φιλόδοξα στα επόμενα, στην επόμενη επιτροπή. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι αυτή η, το μηδενικό όραμα έχουμε, έχει καλυφθεί κατά 60%. Το 40% μπορούμε να το κάνουμε τα επόμενα 30 χρόνια. Και μπορούμε να το κάνουμε γιατί κάναμε πάρα πολλά πράγματα την τελευταία πενταετία. Ελπίζω ότι αυτό θα υλοποιηθεί, αλλά θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν και είμαι βέβαιος ότι οι μεταφορές θα συνεχίσουν να προωθούν αυτό το όραμα του πρασινίσματος ή το όραμα των μηδενικών εκπομπών. Επίσης, να Βοηθήστε τα κράτη-μέλη. Το τέταρτο πακέτο συνδεδομικών μεταφορών που επιτρέπει στα κράτη επιτέλου, να υλοποιήσουν και να παράσχουν τι υποσχεθήσεις δεσμεύσει. Τα κέρδη που έλεγαν ότι θα, ότι θα έπαιρναν. Εμεί αλλάξαμε τους 14.000 σε 1.600 κανόνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ευρωπαϊκή εθνικοί οι μην ξεχνάτε οι σιδηρόδρομοι ήταν τρομερά εθνοκεντρικοί νομοθετικά. Και συνεχίζουμε τα διασυνοριακά έργα που ελπίζω ότι θα επιτρέψουν την πλήρη υλοποίηση της διαλειτουργικότητας σε όλη την Ένωση ε, μέχρι το 2030 στους σιδηροδρόμους. Αλλά και εσείς πρέπει να είστε. Ε, μέσα στο παιχνίδι, όχι εσείς προσωπικά, ε, το κοινοβούλιο. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορέσετε να επηρεάσετε πάρα πολύ τα κράτη. Δουλέψαμε για ένα πολύ και για την ε, ενδοαστική και για τις ενδοαστικές μεταφορές. Πολλές πόλεις, 600 πόλεις έχουν, μετέχουν αυτή τη στιγμή σε προγράμματα από ανθρακοποίησης και καλύτερης χρήσης των καυσίμων. Δεν έχουμε δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φέρνουμε μαζί τις πόλεις, παράδειγμα, τα εργαλεία, μηχανισμοί ε, επιβολής τελών, ε, ε, ε, συγγνώμη, μηχανισμοί φόρτωσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μπορούμε να αυτή τη στιγμή προωθούμε μέτρα για να έχουμε ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ένωση, όχι 5-6 σε, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και θέλουμε να προωθήσει και η Φιλανδική Προεδρία είναι ο υπολογισμός του κόστου. Πώς, πώς ε, υπολογίζεις το κόστος, ποια φόρμουλα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι η προστιθέμενη αξία των λύσεων που προτείνει η Ευρώπη. Και έτσι βοηθάμε και τις πόλεις στην πραγματικότητα και τους πολίτες. Συνάδελφε Ζήλερ, τα τελευταία χρόνια περάσαμε πολλούς ανώμαλους δρόμους, χτυπήσαμε πολλά ε, σασί, αλλά προχωρήσαμε το πακέτο της ε, κινητικότητας. Ξέρω ότι αυτό που θέσατε είναι σημαντικό. Πρέπει να αποφύγουμε για να βελτιώσουμε το πακέτο, να μην έχουμε άνευ αποτελέσματος ε, ε, αγώνες. Παρακαλώ λοιπόν να συνεργαστείτε με το Συμβούλιο κοιτάζοντας τα σημαντικά. Εγώ παίρνω μηνύματα και επιστολές από χώρες και της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης που διαπιστώνουν σιγά σιγά ότι όλοι χρειάζονται το πακέτο αυτό εν τέλει. Αλλά δεν θα ικανοποιήσει τους πάντες. Προφανώς όλοι πρέπει να δώσουν πίσω κάτι. Και η Κομισιόν έκανε παραχωρήσεις, δέχτηκε κάποιες αλλαγές. Δικαιώματα των επιβατών σιδεδρόμων. Συμφωνώ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κάτι που το προχωρά η Φιλανδική Προεδρία. Η Γενική Διεύθυνση MOVE ήδη έχει μπει στην διαδικασία των συζητήσεων για τα δικαιώματα των επιβατών πολλών ειδών συνδυασμένων μεταφορών που έχει όμως και ζητήματα κυρίως ε, κοστολόγησης και πάλι. Περιμένουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Το Τυρόλο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Τρεις-τέσσερις χώρες στην αίθουσα αυτή, βουλευτές μάλλον από τρεις-τέσσερις χώρες, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Και πιστέψτε με, με απασχολεί κάθε εβδομάδα, μην σας κάθε μέρα. Η πρόκληση που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την τελευταία τριετία είναι να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε με όλες τις πλευρές μία κοινή λύση. Φαντάζεστε ότι οι τέσσερις χώρες δεν έχουν την ίδια προσέγγιση στο θέμα αυτό. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αξιολογούμε την πρόταση της Αυστρίας. Σήμερα στείλα μια άλλη επιστολή την προταση της αυστριας σημερα έστειλε μια αλλη επιστολη ζητωντας περισσότερες λεπτομέρειες για να καταλάβουμε καλύτερα τη νέα, πρόταση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε προς τα έξω ένα πιο θετικό μήνυμα. Μία πιθανή λύση που συζητούμε με τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι διόδια, το Brenner Corridor Mount, διόδια, ένα, ένα, το σύστημα διοδίων του Brenner, του διαδρόμου Brenner. Αυτό ε, είναι θέμα συζήτησης, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η ρήπανση του αέρα στην ε, κοιλάδα του Τυρόλου είναι πραγματικά πολύ σοβαρή και δεν έχουμε πραγματικές εναλλακτικές μέχρι να χτιστεί το τούνελ του Μπρένερ. Ε, ε, το 2027 θα τελειώσει. Έχω πάει εκεί πολλές φορές για να τους ε, στηρίξω ηθικά, αλλά αυτά μπορούν να σκάψουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να σκάψουν πάρα πιο γρήγορα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν κάποιες ενδιάμεσες, άμεσες δράσεις για να μειωθεί και η, η ταλαιπωρία των φωτιγών και η ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής. Λοιπόν, πάμε στις ε, εκπομπές ε, στη θάλασσα. Ε, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ένα από τα θέματα που δουλέψαμε ιδιαίτερα συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια. Και βρίσκομαι στην ευτυχή θέση να μπορώ να σας πω ότι συναντηθήκαμε με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ε, συμφωνήσαμε για όλα τα βασικά θέματα, την ψηφιοποίηση, τη ρήπανση, αλλά επίσης και την απλούστευση των κανόνων και ενδεχομένως και το στρατηγικό προσανατολισμό του μέλλοντος. Όσον αφορά την απομάκρυνση του άνθρακα από τις ε, θαλάσσιες εκπομπές. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό ε, για να επιτευχθεί. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ χρειαζόμαστε την δέσμευση των άμεσα ενδιαφερομένων ότι θα αφαιρέσουν τον άνθρακα ε, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα περιορίσουν και γενικότερα τις εκπομπές, τις θαλάσσιες μεταφορές κατά 50% μέχρι το 2050, αλλά κρατηθείτε με την ρήτρα του 2030 θα τεθούν ακόμα πιο φιλόδοξοι στόχοι. Γι' αυτό λοιπόν να μην ξεχνάτε την υπόσχεση που σας έχουν δώσει. Κατά διάρκεια αυτής της θητείας θα πρέπει να ε, εκφράσουν ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους. Τώρα, αρχίζουμε την ε, συγχρηματοδότηση στην αυπήγηση. Είναι ένα νέο εργαλείο και πιέζουμε και για την ψηφιοποίηση, το, η μονοπευθυντική θηρίδα για την Ευρώπη. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και συνεργαζόμαστε με τον IMO, έτσι η μονοπευθυντική θηρίδα να ισχύει και για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές. Η ψηφιοποίηση θα μας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουμε τις διαδρομές και να έχουμε καλύτερο έλεγχο στην κατανάλωση. Και όσον αφορά τα λιμάνια, επιτέλους φαίνεται ότι θα μπορούμε να ελέγξουμε τα ευρωπαϊκά λιμάνια και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ενθαρρύνουμε και τις τρίτες χώρες να ακολουθήσουν και αυτές εκεί δηλαδή όπου θα ελιμενίζονται τα δικά μας τα σκάφη. Πάντως σας λέω, οι εμπλεκόμενοι στην, ε, στις θαλάσσιες μεταφορές έχουν αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και θέλουν να πάνε ακόμα πιο μπροστά ε, γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει και για τις ε, θαλάσσιες ε, μεταφορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βιολέτα Μπίλτς. Ωραία. Λοιπόν, επόμενες ερωτήσεις. Ένα λεπτό όμως, ε, κυρία Μπιλμπάου, σας βλέπω. Ένα λεπτό. Εμπρός. Ευχαριστώ. Αγαπητή Βιολέτα, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για το έργο σας συνολικά. Ξέρω ότι πολλές φορές ένιωσες μόνη, γιατί η ευθύνη ήταν μεγάλη και δεν σε συνόδευσαν πάντα οι διάφορες κυβερνήσεις των χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, εσύ συνέχισες τις προσπάθειες και το Κοινοβούλιο πάντα σε στήριζε. Ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνώ. Ένωση μεταφορών. Πακέτο κινητικότητας. Και εμένα μου έρχονται επιστολές από διάφορους κλάδους οι οποίοι λένε ότι παρόλο που τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς θα τα θέλανε είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν με το πακέτο αυτό με, ε, κινητικότητας από το να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Πώς λοιπόν θα πιστούν οι χώρες μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που θέλει να συνεχίσει ή συζητιέται να ξεκινήσουμε και πάλι από το μηδέν. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό είναι τριμερής διαλογη για να υπάρχει ισορροπία. Διακόπτη Πρόεδρος, τελείωσε το λεπτό σας. Ο κύριος Ντανιέλ Τάντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την Επίτροπο. Ήσασταν ε, σαφέστατοι και για τις διαδικασίες και για τις προθέσεις σας όσον αφορά το πακέτο κινητικότητας και τις συνδυασμένες μεταφορές. Εγώ θα μιλήσω για κάτι άλλο. Από ό,τι κατάλαβα, όλες οι διευθύνσεις ε, πρέπει να υποβάλουν τρεις συγκεκριμένες προτάσεις με τις οποίες θα ασχοληθεί η νέα Επιτροπή. Μήπως λοιπόν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για το ποια από τις τρεις προτάσεις έχει αναλάβει δικιά σας, το δικό σας χαρτοφυλάκιο να προωθήσει εν ώψη της επόμενης θητείας. Παρακαλώ, κύριο Σφαρμπινιού. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, είμαι νέος, νέο μέλος σε αυτήν την Επιτροπή. Βεβαίως ε, έχω διαβάσει λιγάκι ε, αυτές τις λίγες ημέρες που είχα στη διάθεσή μου όλες αυτές τις διατάξεις που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών. Και ε, ακούσαμε βέβαια μόλις πριν από λίγο ότι υπάρχουν κάποια θέματα που είναι απολύτως απαραίτητα για να βελτιωθούν οι μεταφορές και για να βελτιωθεί και το περιβάλλον. Αναφέρομαι στη ρήπανση, στην κλιματική αλλαγή και σε παρεμφερή. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη κυρία Πρόεδρε γιατί εγώ όχι μόνο συμφωνώ αλλά επαυξάνω κιόλας ε, σε αυτά που είπε η κυρία Επίτροπος. Θέλω όμως να κάνω μία παρατήρηση. Ε, θα κάνω έτσι μία πολύ γενική ερώτηση παρατηρώ ότι σήμερα ο τομέας της ενέργειας, ε, η γεωργία αλλά και οι ιδιώτες έχουν περιορίσει τις εκπομπές ε, κατά 20%. Γιατί στον τομέα των μεταφορών ε, επιδεινώνεται το πρόβλημα των εκπομπών. Πού ακριβώς απέτυχε ο τομέας των μεταφορών και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Φλέγκο, παρακαλώ. Πώς το προφέρετε. Πιτσου Κράπακ. Ευχαριστώ πολύ. Σας συγχαίρω κυρία Μπούλτς. Εγώ είμαι νέο μέλος στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θέλω να σας πω ότι ε, όλοι θέλουν να σε ευχαριστήσουν που ήρθατε. Νομίζω ότι ε, έχετε αφήσει πολύ καλά τα προβλήματα για τους επόμενους και έχετε βάλει και πολύ ψηλά τον πύχη. Τώρα, η ερώτησή μου. Το θέμα ίσως ε, να μην αφορά γενικότερα όλους, αλλά ειδικά εσάς. Είπατε ότι οι μεταφορές είναι κινητήρια δύναμη ε, της οικονομίας. Ε, θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πού ακριβώς πρέπει να επενδύσουμε για να έχουμε το μεγαλύτερο κέρδος. Και μην ξεχνάτε, κέρδισα και τρία δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, αλλά με το όνομά σας ακόμα. θα σας ονομάζω έτσι. Ε, κυρία πάρνε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βούλκ, το είπατε εσείς ίδια ότι στην αρχή όταν είχατε έρθει εδώ είχατε ένα διαφορετικό αφήγημα και αλλάξατε. Ε, στην κινητικότητα Προφανώ ε, και πρόκειται για την ευημερία αλλά πρόκειται και για το πώ θα διαφυλάξουμε τον πλανήτη. Βλέπουμε ότι το θέμα του κλίματο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μήπω λοιπόν η επόμενη επιτροπή θα πρέπει να αλλάξει τακτική ε, γιατί ορίζουμε στόχου που πρέπει να βρισκόμαστε στην κινητικότητα μετά από πέντε χρόνια για να επιτύχουμε τους στόχους του Παρισιού και μετά Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τι πρέπει να πετύχουμε στην αστική κινητικότητα, στα περιτά μεγαλεπίβολα προγράμματα όπως είναι οι αυτοκινητιόδρομοι ή άλλα φαραωνικά προγράμματα στους σιδηρόδρομους ε, που δεν ε, θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών. Ίσως λοιπόν επειδή τώρα έχετε την εμπειρία και την ενέργεια έχετε να δώσετε στην επόμενη Επιτροπή συμβουλές έτσι ώστε εκείνη να αρχίσει μεθοδικά πιο σωστά. Ευχαριστούμε κύριε Τεπαρνέ. Ο κύριος Φιντάντσα. Κύριε ε, Πρόεδρε, και εγώ νέος είμαι εδώ, αλλά ε, μέχρι το 2014 ήμουνα σε αυτή την Επιτροπή και έχω συνεργαστεί με τον προκάτοχό σας, τον κύριο Κάλλας, για πάρα πολλά θέματα που βρίσκονται ακόμα στην ημερήσια διάταξη και υπήρχαν ήδη και από παλιά. Θέλω λοιπόν να σας κάνω μία ερώτηση που αφορά σε ένα θέμα για την Ιταλία, αφορά σε ένα στρατηγικό διάδρομο στην Ιταλία έχουμε ακούσει ότι τώρα ένα χρόνο μετά από σκανδαλώδεις ε, καθυστερήσεις η τελική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός εχθές ε, έδωσε το πράσινο φως για την υλοποίηση της ε, διαδρομής το Ρήνο λιον με σιδηρόδρομους ταχείας, υψηλής ταχύτητας. Οι ημερομηνίε έχουν πλησιάσει βέβαια πολύ κοντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση ε, κατά 55%. Θέλω να γνωρίζω τώρα από εσά τι θα γίνει, ε, τι περιμένει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ιταλική κυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Μπόρτζια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, Επίτροπε, και ευχαριστώ που απαντήσατε εν μέρη στο ερώτημά μου. Το Μπρένερ είναι η περιοχή που έχει το μεγαλύ, τη μεγαλύτερη ορία εμπορευμάτων αποτείνεται στην Ιταλία. 9% του ΑΕΠ συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν να μας ενημερώσετε περισσότερο για το πόσο έχουν προχωρήσει οι εργασίες για την κατασκευή του τούνελ βάσης. Δεύτερον, τι άλλα μέτρα υιοθέτησε η Επιτροπή πέρα της αναθεώρησης της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές για να ενθαρρύνει την ενίσχυση και τη χρηματοδότηση της πλατφόρμας, της ε, συνδυασμένης πλατφόρμας και των υποδομών που είναι βασικά εργαλεία για μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη ρύθμιση των ε, ροών. Επίσης, τι κάνατε ή τι προτίθεστε να κάνετε για να μειώσετε το κόστος που επιβαρύνει τους φορείς. Ευχαριστώ. Κύριε Νόβακ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που μπορώ να χαιρετήσω εδώ την Επίτροπο στη γλώσσα μου στα Σλοβένικα και θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για το έργο σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα είμαι επικριτική σήμερα. Θέλω όμως να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Είπατε ότι 49 μέτρα υιοθετήθηκαν κατά τη ε, διάρκεια της θητείας σας. Και εσεί, ποιο από όλου αυτού του φάκελου, ποιο από όλε αυτέ τι νομοθεσίε πιστεύετε ότι βελτίωσε περισσότερο την καθημερινότητα των ε, πολιτών. ποιο είναι ο φάκελο για τον οποίο είσαστε περισσότερο περήφανοι και στον οποίο συνεισφέρατε περισσότερο. Γιατί αυτό ρωτούν οι δημοσιογράφοι ε, συνήθω όταν συναντιόνται μαζί μα. Και τέλος, τι θα συμβουλεύατε την σλοβενική κυβέρνηση για προγράμματα που θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα. Υποδομές σιδηροδρόμων ή κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την ερώτηση. Παρόλο που είπαμε, δεν θα ρωτάμε τώρα για κάθε χώρα τι συμβουλή να δώσει η Επίτροπος. Για την Ευρώπη μιλάμε. Αλλιώς μεταξύ σας για επιμέρους και προτάσεις που έχετε να κάνετε για τη μία την άλλη κυβέρνηση. Ε, κύριε Ολυβιέ, εσεί τώρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μιλάτε για τις μεταφορές, μιλάτε για την οικολογία. Έχετε δίκιο. Είναι απόλυτα θεμητό και ζωτική σημασία μάλιστα να θέλουμε μεταφορές καθαρέ στην Ευρώπη. Όμω, ομολογείτε από μόνοι σα ότι αν σταματήσουν οι μεταφορέ τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Πράγματι, με τις ελεύθερες συναλλαγές, με τον καταναλωτισμό, τον οιλισμό, εννοείται ότι χρειαζόμαστε τις μεταφορές. Ποτέ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Εμείς πιστεύουμε ότι φυσικά και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε καθαρές και αποτελεσματικές μεταφορές, αλλά και πάνω στο μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε υπέρ της τοπικής προσέγγισης. Ένα σύστημα είναι το δικό σας, το οποίο χρειάζεται όλο και περισσότερες μεταφορές, σε αντίθεση με το δικό μας. Κύριε Γκραπίνη, εσείς τώρα ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το έργο σας έχω το θάρρος να πω ε, βασικά ότι ήσασταν ε, από τους πιο, αν όχι και οι πιο διαθέσιμοι επίτροπος απέναντί μας. Επίσης απαντούσατε πάντα στις επιστολές μας. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν συνάδελφοι. Υπήρξαν αποτελέσματα, αλλά υπήρξαν και καθυστερήσει. Ένα όμω από τα καυτά ζητήματα που παραμένει χωρί λύση είναι το πακέτο κινητικότητα. Ρωτάω λοιπόν ειλικρινά, πιστεύετε, ποια πιστεύετε μάλλον ότι είναι η καλύτερη μέθοδος. Δεν μιλάμε εδώ τώρα για πολιτικά συμφέροντα, ομάδες κτλ. Αλλά λέμε ότι από πλευράς τεχνικής το πακέτο αυτό κινητικότητας πώς θα μπορούσε να προχωρήσει καλύτερα για να βρεθεί λύση στον τριμερή διάλογο. Θα έχουμε ε, καλό ανταγωνισμό, τι θα γίνει με τη ρήπανση, τι θα γίνει με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουν ληφθεί υπόψη όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν είμαι 100% ικανοποιημένη, αλλά πείτε μου μπορεί να επιτευχθεί παρετέρω βελτίωση στο πακέτο. Ευχαριστούμε ε, κύριε Λασαντέ. Α, όχι, εσείς δεν θέλετε το λόγο. Καλώς. Ο κύριος Έντσι, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω ε, στο μέλλον ε, το πλαίσιο και η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους επιτρόπους να αναφέρεται σε μια επίγουσα κατάσταση κλιματική ε, και επίσης και επίγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία όταν μιλάμε για τη ρήπανση της ατμόσφαιρας. Όχι να μιλάμε απλώς για κλιματική αλλαγή αλλά για κλιματική κατάρρευση, για χάος και το θέμα της μετανάστευσης που βιώνουμε ως το αποτέλεσμα ε, της ε, άκρη της χρήσης ε, των πόρων, των πρώτων υλών και της κατανάλωσής τους στον πλανήτη μας. Ανησυχώ ιδιαίτερα ε, διότι θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η γλώσσα και το πλαίσιο που χρησιμοποιούμε σε αυτή την αίθουσα. Μα ζητήστε να είμαστε, να είμαστε θαραλέοι και θα είμαι θαραλέος. Γιατί δεν πληρώνουν οι ρηπαίνοντες, τι έγινε με το Dieselgate, γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να ελέγχει τόσο πολύ ε, το Κοινοβούλιο και τις χώρες μας. Δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ θέλω να πω παρακαλώ εκπαιδεύστε τους ηγέτες των χαρών των χωρών μας ε, για να χρησιμοποιούν τη σωστή γλώσσα και έτσι να παρουσιάζουν την επίγουσα κατάσταση που υπάρχει λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστούμε πολύ για τον ενθουσιασμό στην παρέμβασή σας. Παρακαλώ, εσείς τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι υποδομές. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στους βασικούς οδικούς άξονες μέχρι το 2030. Εγώ όμως έχω την εντύπωση ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο τοπικό οδικό δίκτυο, ε, διότι αυτό μην ξεχνάμε ότι δεν είναι πολλές φορές ικανοποιητικό Κατανοώ βέβαια ότι η αρμοδιότητα δεν είναι καθαρά ευρωπαϊκή, αλλά τελικά γιατί ε, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα όπου ε, δεν χρησιμοποιούνται παρκώς οι πόροι που υπάρχουν για να υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το τοπικό δίκτυο. Μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουμε και θα έχουμε πολύ καλό ε, δίκτυο στους βασικούς άξονες. Κυρία Επίτροπε, έχοντας κατά νου τη δική σας την εμπειρία, πιστεύετε ότι ε, μπορείτε να λύσετε αυτό τον φαύλο κύκλο τουλάχιστον κατά, την, ε, κατά το επόμενο Συμβούλιο, την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Υπάρχει ε, αυτό το ο τσακωμός ε, του 5G στράφει κατά των πολιτών. Τελικά πέτυχε η νομική πράξη. Τι θα γίνει τελικά στο μέλλον. Ε, θα καταθέσετε μία πρόταση ουδέτερη προς την τεχνολογία για να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία ή θα το αφήσετε αυτό το θέμα ε, στον ιστή διαδοχό σας. Γιατί αν το κάνετε νομίζω ότι θα αφήσετε τη σφραγίδα σας με αυτό το θέμα για τη θητεία σας. κύριος Νακόφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Αγαπητή Επίτροπε, ευχαριστώ για το έργο σας τα τελευταία πέντε χρόνια. Και χαίρομαι που έχουμε τη συζήτηση αυτή μετά τις εκλογές, γιατί νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να προχωρήσουμε και να λύσουμε το θέμα του πακέτου κινητικότητα. Αν το είχαμε κάνει πριν τι εκλογέ. καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα ήταν άσχημα. Ήλπιζα ότι θα υπάρξει στήριξη και ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλά από τα αμφιλεγόμενα θέματα που περιλαμβάνει το πακέτο κινητικότητας με την ρήπανση που μας έρχεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία μας διχάζουν. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει ένας επικοδομητικός τρόπος για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, το πακέτο κινητικότητας εμποδίζει και άλλους φακέλους στις ιδιασμένες μεταφορές, για παράδειγμα. Ε, παρόλο που εγώ ήμουν εισηγητή και με ιδιαίτερη χαρά δούλεψα πάνω σε αυτό. Οπότε κάνω έκκληση σε όλου του συναδέρφους να βρούμε ένα κοινό τόπο. Τέλο. Μερικέ φορέ έχω την αίσθηση εδώ ότι είμαι μέλο τη επιτροπή περιβάλλοντο. Μα εμείς τις μεταφορές πρέπει να έχουμε υπόψη μα. και όχι αυτό κατά προτεραιότητα, ακόμα και αν έξω έχει 40 βαθμού. Ε, το πακέτο κινητικότητας αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών. Μας αρέσει ή όχι, εδώ δικιά μας αρμοδιότητα είναι. Η κυρία Γκαρσία τώρα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρέμβασή, την παρουσίασή σας και για το έργο σας όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι καινούργια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά για να προχωρήσουμε μαζί σας. Συμφωνούμε όσον αφορά τις καθαρές μεταφορές και την ανησυχία που εκφράζετε κι εσείς για έλλειψη εργαζόμενων οδηγών και για το θέμα της ψηφιοποίησης επίσης ή του αυτοματισμού των οχημάτων Κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια και μας το εξήγησε και η Φιλανδική Προεδρία σήμερα το πρωί ότι θα το βρούμε μπροστά μας όλο και περισσότερο. Οπότε ψηφιοποίηση, αυτοματισμός πρέπει να συνοδεύονται από μια δίκαια μετάβαση και να προβλέπεται χρηματοδότηση και βοήθεια στον κλάδο για να μην χαθεί το εργατικό δυναμικό και για να βελτιωθούν οι γνώσεις τους με θετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μάης, έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το 2015 υπήρξε μία δίωλωση για την ποδηλασία και την ανάγκη η ποδηλασία να αντιμετωπίζεται ως μία μορφή μεταφοράς όπως οι άλλες και οι επενδύσεις σχετικά να αυξηθούν και ταυτόχρονα να αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου κατά 50% μέχρι το 2030. Πέρασε και ένα, ε, βγήκε και ένα ενδιαφέρον κείμενο για την πολιτική υποδηλάτου της Ένωσης. Η ερώτησή μου είναι, τι πρόοδος υπήρξε στον τομέα αυτό, στη στρατηγική για την ποδηλασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε πρόοδος, σοβαρή πρόοδος τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μια ακόμα ερώτηση, ασφάλεια στον δρόμο. Το 2018 είχαμε 26.000 θανάτους στο δρόμο. Τι προθέσεις έχετε για την ασφάλεια στους δρόμους. Ξέρετε, πέρασα το χρόνο μου. Τελευταία ερώτηση. Η αλλαγή του της ώρας, της θερινής ώρας. Αλλά ξέρω ότι δεν θα προλάβω να απαντήσετε σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μέες. Daunting. Um, Clearly you yourself admit that we have a huge... Ευχαριστώ Επίτροπε. Όντως, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση αν θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Αναφέρετε ότι έχετε νέες προτάσεις, αλλά και με τις νέες προτάσεις υπάρχει ένα κενό 40% για να πετύχουμε το όραμα αυτό που θέλετε έχετε κάτι που να μετανιώσατε που δεν κάνατε ή που δεν υλοποιήθηκε. Τι πρέπει να προχωρήσουμε ε, στο μέλλον. Με κάποιο τρόπο πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Επιτροπή ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο κόσμος κινείται, θέλει να κινείται και αυτό δεν θα αλλάξει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ωραία το είπατε το όνομά μου, Καμπονέ ναι, με λένε. Καλωσορίσατε κύριε Μπούλτ. Συμφωνώ με αυτά που αναφέρθηκαν πριν από μένα. Χαίρομαι που η Ιταλική κυβέρνηση έδωσε το τελικό OK στη διαδικασία του τρένου υψηλή ταχύτητας στο Ρήνο Λιόν. Δεν είναι σημαντικό μόνο το έργο αυτό καθεαυτό και για τις εμπλεκόμενες περιοχές και με το Connecting Europe Facility θα έπρεπε να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με έργα στρατηγικής σημασίας που θα αφορούν τις παραμεθόριε περιοχέ. Εγώ είμαι από τη Γένοβα, δεν θέλω να μιλήσω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είμαι από μια πόλη όπου συνέβη η κατάρρευση του, της γέφυρας Μωράντη στη Τζένοβα πέρσι. Δύο σημαντικά ζητήματα λοιπόν. Ασφάλεια των υποδομών αφενός. Πρέπει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, ένα έργο που θα ασχολείται με τον έλεγχο και την επαλήθευση του, του, της ποιότητας των υποδομών, μεγάλων υποδομών με τις οποίες ε, ε, που μας απασχολούν τώρα για το μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη ως δίδαγμα της τραγωδίας στη Γένοβα. Ευχαριστώ. Κύριε Αμπούλτς, έχετε 22 ερωτήσεις μόνο, εντάξει. Και 13 λεπτά. 47 δευτερόλεπτα να ερώτηση δηλαδή έχετε. Όλες οι ερωτήσεις που θες είναι σημαντικές. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω λεπτομεριακά σε όλες. Ή θέλαμε μετά τις διακοπές σας να σας στείλουμε ένα fact sheet ε, με ό,τι πετύχαμε, τις εκκρεμότητες και ποιους τομείς θεωρούμε ως ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί τα επόμενα, στην επόμενη φάση. Αυτό θα το πάρετε όλοι σας λοιπόν. Να απαντήσω σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν και που μπορούμε να τους δούμε στο συνολικό πλαίσιο. Α, τα, τα, τα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Υπάρχουν προτάσεις διεύρυνσής τους και επέκτασής τους. Θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση και το 2020 θα έχουμε τις προτάσεις για την πιθανή επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ε, διευρωπαϊκών μεταφορών. Αλλά προσέξτε, η έμφαση, ε, η προτεραιότητα και η αρμοδιότητα είναι των κρατών μελών. Ε, εμείς έχουμε το συντονισμό μετά την ε, μελέτη αντικτύπου των προτάσεων που θα τεθούν επιτάπτως θα προτείνουμε με βάση τα κριτήρια που είναι γνωστά ο κατάλογος βέβαια τον κατάλογο των μελλοντικών συνεπενδύσεων. Τώρα το Λιόν Τωρίνο και κάποια άλλα μεγάλα έργα που αναφέρονται η, πρώτη, η βασική απόφαση ανήκει στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προτείνουν και αν προτείνουν και πιστεύουν ότι κάποια έργα είναι αναγκαία, εμείς ξαναβλέπουμε με βάση τα κοινά κριτήρια τις προτάσεις, απαντούμε στις ανάγκες και απαντούμε στις ανάγκες που εκφράζονται. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε την ομιλία του Ιταλού Πρωθυπουργού που βεβαίωσε ότι υποστηρίζει το έργο το Τωρίνο, αλλά περιμένω την επίσημη ε, επιβεβαίωση εγγράφος για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτήματα για την ε, αποτελεσματικότητα και την απο, αφαίρεση του άνθρακα, την μετατροπή των ευρωπαϊκών μεταφορών σε μη ε, μεταφορές ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο έχουμε αρνητικές εξωτερικές δαπάνες από τις μεταφορές. Σας δώσαμε μία έκθεση που δείχνει ανακράτους μέλος και αναμορφή μεταφοράς ποιος συμβάλλει με πόσο. Με βάση αυτό πιστεύω αποφασιστικά ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα οικονομικά προς όφελος αυτών των μέσων μεταφοράς που δεν ε, που δεν ε, ρηπαίνουν. Εσωτερικές πλωτές μεταφορές, θάλασσα, τρένο. Το 60% της ρήπανσης είναι από τις οδικές και το 16% από αυτά ε, είναι από τα γιοταχή. Και εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε και συνδυασμένες επιβατικές ε, συνδρομικές μεταφορές. Αλλά αυτό πρέπει να προταθεί. Δεν μπορούμε να χτίσουμε εμεί ω Κομισιόν ε, να κατασκευάσουμε ε, γραμμές ιδιοδρόμων ή να παράσχουμε υπηρεσίες. Το προσπαθούμε με τις συνεπενδύσεις. Αυτό προσπαθήσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια και αυξήσαμε σημαντικά την, ε, τις επενδύσεις, τις ε, μεταφορές στην Ευρώπη τα τελευταία 4,5 χρόνια. 200 δις. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά χρειαζόμαστε έργα. Οι, οι επενδυτές ενδιαφέρονται διότι έχουν μία Έχουμε μια στρατηγικά σαφή ημερήσια διάταξη, διαφάνεια, προβλεψιμότητα, δεσμεύσει, αλλά χρειαζόμαστε καλά σχέδια, καλά project. Και αν με ρωτήσετε πού να επενδύσω, σα πω. Πολύ, πολύ ε, ε, συνδυασμένη χρήση, ε, με, κέντρα φόρτωσης, ε, πολυ, ε, συνδυασμένες μεταφορές στο εσωτερικό των πόλεων, όπου μπορεί εύκολο ο επιβάτης να περάσει από τον ένα στον άλλο τρόπο μεταφοράς και τελικά να εξασφαλίσουμε ότι οι περισσότερες ε, μεγά, μακράς απόστασης μεταφορές στην Ευρώπη πηγαίνουν είτε συνδρομικά είτε από εσωτερικές πλωτές οδούς. Αλλά οι προκλήσεις που υπάρχουν και μας το λένε είναι το εξή. Μας το λένε οι φορείς. Ε, δεν είναι αξιόπιστα τα τρένα. Υπάρχουν τρύπε. Ε, και αυτό και προτιμούν την, καλή, την επιλογή που αποδίδει για αυτούς, το, αυτοκίνητο, το φορτηγό. Προχωράνε και τα ΣΥ και οι αλλά προχωράνε αργά. Γι' αυτό θέλουμε να υλοποιήσουμε το τέταρτο συνδρομικό πακέτο το συντομότερο δυνατό. Γιατί κάνει αυτό που θέλουμε. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τη ρήπανση. Είμαστε επίσης υπέρ του τρένου υψηλή ταχύτητα. Θέλουμε το 2030 να συνδέεται όλη η Ευρώπη με κλασικό σιδηροδρόμο, δηλαδή έως 220 χιλιόμετρα την ώρα. Ταυτόχρονα όμως παροτρύνουμε την κατασκευή τρένων υψηλής ταχύτητας, εκεί που είναι τα κέρδη, στο Eurostar για παράδειγμα, Όπω ξέρετε το Eurostar ε, πήγε, επέξέτεινε τι υπηρεσίε του, πήγε στο Άμστερνταμ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ένα τέτοιο τρένο να συνδέει όλες τις πρωτεύουσε ή τις μεγάλες πόλεις Ευρώπης. 500-600 χιλιόμετρα ε, το τρένο είναι καλύτερη επαρκής λύση. Αλλά κανεί δεν τολμά να το κάνει. Βλέπουμε όμω ότι υπάρχουν βελτιώσεις. όσο πιέζουμε, όσο δίνουμε κίνητρα, προχωράμε. Βοηθήστε μα να το περάσουμε αυτό. Η Κομισιόν είναι έτοιμη, δεν είναι εμπόδιο εδώ. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε να συνδέσουμε την Ένωση. Γιατί αυξάνεται η ρήπανση, γιατί ξεκίνησε να λειτουργεί η ενιαία αγορά. Ο κόσμος συνδέεται, δουλεύει ε, και ε, κεφαλαιοποιούμε από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς, αλλά γίνεται μεγαλύτερη ε, κινητικότητα στην Ένωση. Και αν δεν προχωρήσουμε στην, στις μηδενικές εκπομπές θα συνεχίσει να αυξάνεται η λίπανση. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει την απλοποίηση των επενδύσεων, ούτως ώστε των επενδύσεων που έχουμε συμφωνήσει από κοινού, ώστε να ξεπεραστούν γρήγορα οι διοικητικέ διαδικασίες. Όχι, να, όχι 3 και 5 και 10 χρόνια. 10 χρόνια θέλει μερικέ φορέ να προχωρήσουν τα έργα. Και το άλλο είναι η εφαρμογή των μεγάλων υποδομών που θέλουν 7 με 15 χρόνια. Γι' αυτό είναι σημαντικό ένα στρατηγικό προγραμματισμό. Ένα δρόμο μπορεί να το κάνει πιο γρήγορα, αλλά πολύ πιο αργά. Θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για να κάνει γέφυρε, σιδεροδρόμου και τέτοια. Αυτές οι στρατηγικές πρέπει λοιπόν να περνάνε μέσα από πολλές θητείες και άρα πρέπει κληρονόμησα πολλά έργα, έργα υποδομών από τον κύριο Κάλλα, τον προκατοχό μου και προφανώς και ο διάδοχός μου θα έχει πολλά δικά μου. Άλλο θέμα ο Ριπένον πληρώνει. Αλλά εδώ είναι θέμα πολιτικής απόψεως. Ποιο θα πληρώνει. Η κοινωνία, η φύση, ο Ριπένον. Αυτή είναι μια σκληρή συζήτηση όχι μόνο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά και στην Επιτροπή Μεταφορών γιατί έχει σχέση με την Επιτροπή Μεταφορών. Πράγματι στις μεταφορές πρέπει να περάσουν νέα μηνύματα. Ίσως να έχετε δει ότι έχουμε ήδη σαγάγει οριζόντιες προτεραιότητες, έξι οριζόντιες προτεραιότητες για αυτή τη θητεία ρήπανση, απομάκρυνση του άνθρακα, ε, ψηφιοποίηση και κατόπιν καινοτομία, ε, κινητικότητα, διότι αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τους ανθρώπους και παγκόσμια ηγετική θέση και επενδύσεις. Όλα αυτά για να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας. Ε, την ε, διαχείριση των εξωτερικών παραγόντων ε, πλησιάζοντας το μηδέν, βελτίωση της αποδοτικότητας ε, και τρίτον βελτίωση της διασύνδεσης μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο μοντέλο στις μεταφορές θα είναι ψηφιακό και επιτρέψτε μου σύντομα να απαντήσω και στην πρόκληση CITS. Βεβαίως και είμαι ε, απογοητευμένη με αυτά που συνέβησαν, με όλες αυτές τις δραστηριότητες των λόμπις, ε, πολύ άδικες ε, και δεν εξήγησαν τα επιτεύγματα, τους στόχους, τα μέσα, πώς η Επιτροπή επιθυμεί να εφαρμόσει το CITS. Και στο τέλος το Συμβούλιο δεν αναχέτησε την εφαρμογή αυτής της κατεξουσιοδότηση πράξης ε, λόγω του 5G, ε, αλλά ε, υπήρξαν κάποια νομικά θέματα νομικής φύσεως που προβλήθηκαν και εντάξει σας το λέω, τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα νομικής φύσεως θέματα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το CITS ε, θα μπορούμε να το διατηρήσουμε όπως έχει προταθεί και θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι όσον αφορά το 5G Πρόκειται για ασφάλεια, να ε, σώζονται ζωές, οι μεταφορές να είναι πιο αποτελεσματικές, να αφαιρεθεί ε, ο ανθρώπινος παράγων ε, που δεν επιτρέπει να αντιδράσει κανείς γρήγορα σε ορισμένες περιπτώσεις. Και δεν είναι υπηρεσία, είναι μια λειτουργία, είναι ένα σύστημα που επιτρέπει να μεταφέρονται πληροφορίες για το τι ακριβώς γίνονται γύρω σου όταν οδηγείς. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η βιομηχανία θα το χρησιμοποιήσει και θα συνεχιστεί η πίεση από την αγορά και παράλληλα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους ε, ενδιαφερόμενους και να βελτιώσουμε αυτό που πρέπει να βελτιωθεί. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για ανταγωνισμό με το σύστημα 5G. Ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα θα περάσει και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε τους στόχους. Και κάτι άλλο, το οποίο ε, θα το δείτε πολύ συχνά ε, να σας απασχολεί, η κινητικότητα ως υπηρεσία. Με τα, τα διάφορα που υπάρχουν, ε, σύστημα πληροφόρησης για τις εσωτερικούς δρόμους, τους πλωτούς. Αν προχωρήσει το πακέτο της κινητικότητας και εκεί θα υπάρχουν εξελίσεις. Κατόπιν υπάρχουν τα θεμέλια για την χρήση ε, ψηφιακών λύσεων. Οι εφαρμογές μπορούν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στα κινητά συστήματα. Θα μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ε, στην επιμελητία, αλλά και πολλές άλλες ε, πολυτροπικές λύσεις για συνδυασμένες μεταφορές. Νομίζω όλα αυτά θα τα εξηγήσετε, αλλά σας παρακαλώ να προσέξετε πάρα πολύ σε κάτι το οποίο, με το οποίο θα πρέπει να συνεργαστείτε και με τον ανταγωνισμό, δηλαδή την κακή χρήση των νέων τεχνολογιών. Με τα blockchains, πολύ ενδιαφέρον αυτό ε, και υπάρχει στις μεταφορές, αλλά μέσω αυτού είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν κλειστά οικοσυστήματα και μονοπόλια. Αλλά πρέπει να έχουμε τις σωστές ε, εφαρμογές, τα σωστά ε, interfaces για να στηρίξουμε το μοντέλο του ανταγωνισμού. Δυστυχώς δεν, δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Αν χρειαστεί θα επανέλθω ε, γραπτά για να απαντήσω και άλλες ερωτήσεις που θα θέσετε κυρίως για το πακέτο της κινητικότητας. Νομίζω ότι το πακέτο αυτό είναι πολύ καλά προετοιμασμένο. Βεβαίως ε, δεν είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για βελτίωση διότι παρότι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου βρίσκονται πολύ κοντά, μόλις είναι έτοιμο το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα εφαρμόσει και εάν υπάρχει βούληση ε, των συντονιστών και στις δύο πλευρές ε, θα προχωρήσουμε γιατί υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Και τέλος ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για την εξαιρετική Προεδρία και τα πήγε τόσο καλά που να, ξαναβρίσκεται εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι αποτελεσματική ε, για να ε, λειτουργήσουν τα δύσκολα θέματα, να υπάρχει διάλογος με την Κομισιόν και, με τα κράτη-μέλη και ε, προσβλέπω στους πολύ καλούς συντονιστές εναποκείται πλέον σε εσά ε, για να βρείτε τους σωστούς δρόμους προς τα εμπρός. Ήταν τιμή και χαρά για μένα το ότι ε, μπόρεσα να συνεργαστώ με σας, με τους Ευρωπαίους πολίτες και νομίζω ανεξάρτητα που θα ξανασυναντηθούμε θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ και ε, καλή τύχη στα μελλοντικά σας προγράμματα. Κύριε Βιολέτα Μπούλτ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά μα μιλάτε σαν να έχει τελειώσει η δουλειά. Δεν έχει τελειώσει. Μα μένουν πολλέ διαπραγματεύσει ακόμα. Και εμεί είμαστε έτοιμοι για τι διαπραγματεύσει. Και μη φεύγετε, γιατί έχουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη τώρα. και πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά. Οπότε αν θέλετε να φύγετε από την αίθουσα να φύγετε ήσυχα, αλλιώς είμαστε στο σημείο 4. Λέει πρόεδρος. Αν θέλετε να βγείτε από την αίθουσα ήσυχο. Το σημείο 4. Οι σοσιαλιστές εκεί, οι διάφοροι σύμβουλοι, παρακαλώ, ήσυχα. Αν θέλετε ε, να μιλάτε μεταξύ σας, εκτός εθούσης παρακαλώ. Βίκτορ, εκτός. Συνεχίζουμε. Σημείο 4, πολύ βασικό για την Επιτροπή μας. Πρόκειται για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, όλα τα τμήματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν την δημοσιονομική διαδικασία για το 2020, Προϋπολογισμός 2020. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για το τελευταίο χρόνο της περίοδου του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου που έχουμε τώρα και πρόκειται για τον προϋπολογισμό, τον τελευταίο που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή Γιούνκερ. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντάνιελ Φρόιτ και μετά θα δώσω το λόγο στους εισηγητές και μετά θα σας παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Φρόιτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούσαμε σήμερα ότι 25% είναι υπεύθυνε οι μεταφορές για τα... τις εκπομπές από του θερμοκηπίου. Και έχουμε δει και σε άλλου τομεί ότι τα τελευταία χρόνια μειώνονται οι μεταφορές, η, η Μόνο στι μεταφορές δεν μειώνεται η ρήπανση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε περισσότερα οχήματα στους δρόμους μας, και έτσι έχουμε περισσότερε εκπομπέ. Όλε οι χώρε μέλη πάντω έχουν ε, συνυπογράψει τη Συμφωνία των Παρισίων και τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η εκλεγμένη πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μείωση μέχρι το 2050 ουδετερότητα όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο καθήκον. Πώς θα πετύχουμε αυτήν την ουδετερότητα στις μεταφορές μέχρι το 2050. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμεθα και πρέπει να αρχίσουμε τώρα να το κάνουμε αυτό. Γιατί κυρίως όταν μιλάμε για σχέδια μεγάλων υποδομών όπως είναι το τούνελ του Μπρένερ ή για άλλο εξαπλισμό, αυτά τα πράγματα κρατάνε δεκαετίες. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Όταν λοιπόν κοιτάω τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και τους στόχους που έχουμε θέσει με τη Συμφωνία των Παρισίων, πρέπει να πω ότι ο προπολογισμό του 2020 για τις μεταφορές δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είτε λοιπόν μπαίνουμε σε ένα σενάριο όπου μεγάλα τμήματα του πλανήτη μας δεν θα κατοικούνται πια, δεν θα μπορούμε να τα κατοικήσουμε ή αλλιώς θα πρέπει να σταματήσουμε την κινητικότητα και τις μεταφορές οι οποίες οδηγούν σε περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κάτι το οποίο βέβαια θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μετακινόμαστε και την οικονομία μας. Παρά λοιπόν τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, το Συμβούλιο θέλει να περικόψει τον προπολογισμό που ήδη είναι περιορισμένος για τις μεταφορές. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλύτερες συνδρομικές ε, συγκοινωνίες, συνδέσεις μεταξύ των χωρών μελών. 1,5 δισεκατομμύρια ετησίως αλλά νομίζω ότι μόνο μια κυκλοφορική συμφόρεση ε, το χρόνο θα γλιτώσουμε. Από το Βέλγιο να πάει κάνει στο Άχεν, για παράδειγμα, που είναι δικιά μου η πόλη, σίγουρα χρειάζεται τουλάχιστον αυτό τον προπολογισμό, αν και όχι παραπάνω, που προβλέπεται για ολόκληρη την Ήπειρο. Συνεπώς, πρέπει να ξαναδούμε τη χρηματοδότηση των μεταφορών. Οι διατάξει που έχουμε για το κλίμα, το InvestEU, πρέπει να αποτελέσει και το κριτήριο για την χρηματοδότηση των μεταφορών. Η μερική συμφωνία που έχουμε για το InvestEU λέει ότι σχέδια τα οποία συνάδουν με τους στόχους για το κλίμα μόνο θα επιλέγονται, αλλιώς όχι. Και πάντα θα υπάρχει το κριτήριο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Όντως αυτή πρέπει να είναι και η βάση για κάθε χρηματοδότηση με την οποία θα συμφωνήσουμε. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι όταν πρόκειται για τις επενδύσεις, στις ε, υποδομές μεταφορών, ο σιδηρόδρομος και η βιώσιμη κινητικότητα πρέπει να αποτελέσουν την προτεραιότητά μας και να ενισχύσουμε βέβαια και τις υποδομές ασφάλειας ε, στις μεταφορές. Πολλοί θάνατοι ή δυστυχήματα έχουν σαν θύματα πεζούς ή ποδηλάτες. Το 2020 επίσης είναι το έτος αναθεώρησης της εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και θέλω λοιπόν να ζητήσω να λάβει υπόψη της όλα αυτά τα κριτήρια στην διαδικασία αναθεώρησης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν βέβαια κάνει κάποια πρόοδο όσον αφορά τη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, όλα αυτά η συμμετοχή των ε, πολιτών στα σχέδια αυτά πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό προτείνω ένα σχέδιο το οποίο έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στο στα περιφερειακά ταμεία και θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο εργαλείο και για τη συμμετοχή των πολιτών ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και στον τομέα των μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στα σχόλια των συναδέρφων. Ευχαριστώ. Κύριε Τέλερ, έχετε το λόγο μια και δεν μπορεί να είναι εδώ ο κύριος Μαρινέσκου. Για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, το σχέδιο προϋπολογισμού του 20 με την περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων 5 εκατομμύρια για την κοινωτικότητα μεταφορών και 3 εκατομμύρια για τις ε, πιστώσεις που μπορούν να επιτρέψουν ε, την αύξηση του ποσού. Ο κύριος Μαρινέσκους και ο δισηγητής θα υποβάλει δύο κατηγορίες τροπολογιών για τα πιλωτικά σχέδια και τα, ε, για τις τροπολογίες για τα TEN στο πακέτο 6 θα επαναφέρει τα ποσά όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις οποίες, το οποίο περιέκοψε το Συμβούλιο επίσης θα αυξήσει τα ποσά για την ε, ημερήσια διάταξη ευρωπαϊκών αερομεταφορών από 37,9 σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα εξετάσουμε πιο προσεκτικά την γνωμοδότηση του προϋπολογισμού και θα την αλλάξουμε χρειαστεί το Σεπτέμβριο. Κυρία Γκραπίνη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτό παραπέμπει στην προηγούμενη συζήτηση, ο βασικός, ε, το βασικό προπολογισμό για τις μεταφορές. Γι' αυτό δεν ξέρω γιατί το Συμβούλιο πρότεινε περικοπές σε κάποιους τομείς. Ως εισηγήτρια, ως εισηγήτρια για τους σοσιαλιστές θα υποβάλω προτάσεις για να αποκαταστήσω το επίπεδο του προπολογισμού στο προγενέστερο επίπεδο. Είναι σαφές ότι υπάρχουν μεγάλες δημοσιονομικές αποκλήσεις, το ανέφερε και συνάδελφος από το ΕΛΚ, για την 060204 θέση υπάρχουν αποκλήσεις, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Μεταφορών, κατόπιν υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις και αλλού, παραδείγματος χάνει στις Είναι σαφές ότι ο προπολογισμό που προετοίμασε η Επιτροπή δεν είναι ιδεώδης. Τώρα που μπήκε για το Συμβούλιο και κάνει και περαιτέρω προ, προ, ε, αυτό δεν στέκει. Θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες σχετικά. Κύριε Μποζαντίας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κι εγώ ένα λεπτό έχω, πρόεδρε. Δύο-τρία σημεία. Πρώτον, ποιοι είναι οι στόχοι σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Πρέπει να συνεχίσουμε με τα προγράμματα και έργα ΣΒΙΤ που υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Πέρυσι το τελευταίο δημοσιονομικό έτος είναι κρίσιμο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και συνέχεια των υφιστάμενων έργων και να καθορίσουμε τις κομβικές προτεραιότητές μας. Τώρα για, την, για τα πιλωτικά σχέδια θα πρέπει να έχουμε ως στόχο τα αποτελέσματα και να αναζητήσουμε της, ε, προς την προστιθέμενη αξία της Ένωσης. Τουρισμός, άλλη προτεραιότητα. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ε, του τουρισμού ειδικό. που θα εξετάζει τον αντίκτυπο οικονομικό και κοινωνικό. Κλείνω. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τις την υπηρεσία μεταφορών, τις υπηρεσίες μεταφορών της Ένωσης για τη δουλειά που έχουν κάνει. Έχουν κάνει πραγματικά σημαντική, ε, έχουν συμβάλει σημαντικά στην διαμόρφωση των θέσεων της Ένωσης. Αυτά. Ευχαριστώ. Είδε. Κύριε Ζήλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το ECR ε, πάντα στηρίζει την θέσπιση ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού. Για μας είναι πολύ σημαντικό πώς δεπανώνται τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά ε, πιστεύουμε ε, το ECR στηρίζει αυτά που είχαν προβλεφθεί αρχικά στον προπολογισμό στις περισσότερες γραμμές. Βεβαίως, ε, καθαρά πολιτικά, ε, θέλω να πω ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν ε, τα μεγαλεπίβολα έργα Connecting Europe Facility και αυτό το σύστημα ανάμιξης το οποίο ε, προέκυψε τα τελευταία χρόνια για τις ε, γραμμές του προεπλογισμού. Είμαστε ε, φυλακτικοί για τα πιλωτικά προγράμματα, τις προκατακτικές δράσεις γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις εκεί που υπήρξαν δεν βοήθησαν να υπάρχει σημαντική πρόοδος. Προσβλέπουμε στο σχέδιο της γνωμοδότησης και θα καταθέσουμε κάποιες μικρές τροπολογίες σε κάποιες γραμμές. Κύριε Κουντουρά, παρακαλώ. Η πολιτική μεταφορών της Ένωσης είναι κεντρικής ε, σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και από τις μεταφορές εξαρτώνται ορισμένες από τις θεμελιώδεις πολιτικές της Ένωσης. Η ενιαία αγορά με την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών και η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές κατακτήσεις. Η πολιτική αυτή λοιπόν έχει ανάγκη από ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό όχι μόνο για να ολοκληρώσει τους βασικούς διαδρόμους μεταφορών αλλά και για να αντιμετωπίσει μία επίγουσα κρίση την κλιματική αλλαγή. Τη διτή αυτή λοιπόν πρόκληση πρέπει να έχουμε υπόψη όταν συζητάμε στην Επιτροπή αυτή για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ και στη σημασία των πιλωτικών προγραμμάτων για την Επιτροπή μας λήψη γραμμή για τον προπολογισμό για τον τουρισμό στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο μας παρέχουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την περιορισμένη αλλά αναγκαία χρηματοδότηση δράσεων στον τουρισμό και είναι ίσως μια απτή απόδειξη ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και πρέπει να αναβαθμιστεί άμεσα και να έχει βέβαια τη δική της ε, γραμμή προϋπολογισμού. Ένα παράδειγμα είναι το πιλωτικό πρόγραμμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της κουραζιέρας που μπορεί να οδηγήσει πολλές περιοχές σε ορθότερη διαχείριση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Δυστυχώ όμω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα το σχετικό διαγωνισμό με κίνδυνο να χαθεί η χρονιά και είμαι πεπισμένη ότι δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό κίνητρο πίσω από αυτή την καθυστέρηση. Είναι όμως σημαντικό για μας τους ευρωβουλευτές που προτείνουμε αυτού του είδους τα προγράμματα να μπορούμε να εμπιστευτούμε την Επιτροπή και την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Μπιλμπάου, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι απαράδεκτη αυτή η μείωση που προτείνει το Συμβούλιο στον προπολογισμό. Εμείς έχουμε συγκεκριμένους στόχους, κλίμα, ψηφοποίηση, αυτοματισμός κλπ. κλπ. Πώς δεν τα κάνουμε όλα αυτά. Αν το Συμβούλιο θέλει μείωση του προπολογισμού, πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να είμαστε απόλυτοι και μόνο θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας αν τα σχέδιά μας έχουν προστιθέμενη αξία. Πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι δυνατόν, όπως ακούσαμε και την Επίτροπο, συνδυασμένες μεταφορές, ε, αποτελεσματικότητα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Συνεπώς, πρέπει να επιμείνουμε. Όσον αφορά τον τουρισμό τώρα, ναι, η Task Force στην προηγούμενη θητεία δούλεψε ώστε ο τουρισμός να έχει ειδική μνήα. Αλλά και πάλι είμαστε θύματα των χωρών μελών που βάζουν την επικουρικότητα και δεν θέλουν να μπούμε σε αυτά τα ζητήματα. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να ξεμπερδέψουμε σε αυτή τη θητεία με αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Είναι ξεκάθαρο. Ο προπολογισμό αυτός δεν είναι δυνατόν να περικοπεί όπως ζητάει το Συμβούλιο. Και γι' αυτό ακριβώς Εμεί θα διατηρήσουμε τον προπολογισμό ω έχει. Αλλά πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι. Έτσι. Υπεύθυνοι. Και όπως πολύ καλά το είπε και ο συγητή, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας. Η πρόταση των πιλωτικών προγραμμάτων είναι ένα θέμα το οποίο συνάδει με τις προσδοκίες των πολιτών. Η κινητικότητα στην καθημερινή βάση, η εγκύτητα Αυτά είναι θέματα που πρέπει να προχωρήσουμε. Και όταν ακούω για τα νυχτερινά τρένα, αυτό πρέπει να είναι πιλωτικό σχέδιο της Επιτροπής μας. Η Αυστρία το έχει εφαρμόσει αυτό με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η Σουηδία επίσης. Είναι κάτι που πραγματικά ζητάνε οι πολίτες. Οπότε κύριε Σιγητά, περιμένουμε να μας Εξηγήστε περισσότερο για το πώς ακριβώς θα συνδυάσουμε το σχέδιό μας με τις προσδοκίες των ε, πολιτών. Λοιπόν, πολλές ήταν οι προτάσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Για να δούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Εσκλατές είναι εδώ. Εδώ είσαστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι εδώ, αλλά συνάδελφος η κυρία Μοτανιά θα απαντήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλωσορίζουμε και εμείς τους νέους ευρωβουλευτές. Ένα πράγμα θέλω να τονίσω που πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με πολλές από τις παρεμβάσεις σας. Θέλω δηλαδή να υπενθυμίσω ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ετοιμάσαμε αυτό το προπολογισμό για το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοείται ότι μένει στο αρχικό ποσό γιατί θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, κυρίως για τη διευκόλυνση για την Ευρώπη. Και υπενθυμίζω επίσης ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Δηλαδή, λαμβάνει υπόψη το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο τη διακυμάθηση κάθε χρόνο και το είχαμε προβλέψει από την αρχή γιατί ξέρουμε ότι τα προγράμματα παίρνουν χρόνο και θέλαμε να προβλέψουμε αρκετά χρήματα στο τέλος της περίοδου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην απειλήσουμε τα προγράμματα με μείωση του προπολογισμού. Τώρα, αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει. Για το χρονοδιάγραμμα, Προσθέτω ότι βεβαίως περιμένουμε την παγιωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, στον και μετά στη συνδιαλλαγή, συγγνώμη, στη συνδιαλλαγή τον Νοέμβριο, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προπολογισμό 2020. σε ευχαριστούμε. Ο εισηγητής, έχετε και πάλι το λόγο για να προσπαθήσετε να απαντήσετε στους κοιόδης εισηγητές να δούμε τι συμπέρασμα βγάζετε, δεδομένο και των προθεσμιών, έτσι. Η έκθεση Ντανιέλ Φρόιτ έχει προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών είναι 26 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Έχετε το λόγο κύριε Φρόιτ. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που είπατε. Βεβαίω και θα σεβαστούμε τις ε, καταληκτικές ημερομηνίε. Αν έχετε ερωτήσεις, οτιδήποτε, η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Με πολύ μεγάλη μου χαρά να συζητήσουμε για όλα αυτά που και μόλις τώρα θίξαμε. Ευχαριστώ. Τροπολογίε πρέπει να κατεθούν μέχρι τις 26 Ιουλίου. Η συζήτηση για την έκθεση θα γίνει ήδη την πρώτη εβδομένα. Κύριε Σιγητά, σας προτείνω σχεδόν να καλέσετε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να έχουμε και μία συζήτηση με βάση τους στόχους που έχετε θέσει. Πρόταση είναι αυτή για να μπορέσει η γραμματεία να το οργανώσει και για να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΤΕΠ. Εάν το δεχτείτε θα φροντίσω να διαμορφώσουμε σχετικά τη μερίσια διάταξη. Συνάδελφοι, λυπάμαι για σας, αλλά δεν θα με ξαναδείτε. Δεν έχουμε άλλο θέμα στην μερίσια διάταξη. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει 3 το απόγευμα 2 Σεπτεμβρίου, 3 με 6.30 και 3 Σεπτεμβρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Να σας ευχηθώ σε όλους. Πολύ καλές διακοπές. Να ξεκουραστείτε. να δείτε και κάποια πράγματα, αλλά κυρίως να φροντίσετε να σας επιτρέψουν να ξανάρθετε πίσω σε φόρμα. Γυρίζοντας, δυστυχώς δεν θα έρθουμε με τρένο υψηλής ταχύτητας, αλλά με τον με ένα αργό τρένο γεμάτο δουλειά, δε, γεμάτο ευθύνες, γεμάτο φακέλους. Καλές διακοπές λοιπόν. Καλές διακοπές και η γραμματεία καλές διακοπές. Ευχαριστούμε όλους για τις για τη δουλειά που έκανε. Ευχαριστεί και τους γερμηνείς η Πρόεδρος. Καλές διακοπές. Τέλος συνεδρίασης.